Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση. Είναι η τελευταία συζήτηση που είχαμε με Πρωθυπουργό ε, στις, στις διαδικασίες αυτές που έχουμε ακολουθήσει, η συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης. Νομίζω ότι η συζητήσεις αυτές ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσες για όλους μας, γιατί ως ευρωβουλευτές πρέπει να είμαστε στην αιχμή του δόρατος ε, όσον αφορά στο μέλλον της Ευρώπης τα αποτελέσματα αυτής, αυτών των συζητήσεων θα τα παρουσιάσω στις 9 Μαΐου, στο επόμενο Συμβούλιο Κορυφής ε, στη Ρουμανία και δράτω με τις ευκαιρίες για να ευχαριστήσω όλους τους βουλευτές που συμμετείχαν σε αυτές τις ε, συζητήσεις. Τις έκαναν πολύ πιο ζωντανές ε, από ό,τι συνηθίζεται. Νομίζω ότι ήταν μια πολύ θετική πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μπορέσαμε να καταδείξουμε ότι το Κοινοβούλιο είναι πραγματικά η καρδιά της δημοκρατίας. Ευχαριστώ για άλλη μια φορά όλους. Ε, καλή προεκλογική εκστρατεία σας εύχομαι και καλό Πάσχα. Λοιπόν, συνάδελφοι, πριν ε, προχωρήσουμε, έχω να κάνω μία ανακοίνωση ότι ο κύριος Ντέβιτ ε, Μπορέλη ε, θα προσχωρήσει στην ομάδα των φιλελευθέρων από τις 17 Απριλίου του 2019. Θα φύγει από τους μη εγγεγραμμένους και θα προσχωρήσει στους φιλελεύθερους. Τώρα λοιπόν προχωράμε με την ψηφοφορία. Το πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη Βλέπω ότι ο κ. Μπιουτικόφερ ζητάει το λόγο. Διαδικαστικό είπατε κ. Μπιουτικόφερ. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Άρθρα 1 και 115 του κανονισμού μας αναφέρομαι σε αυτά και θα ήθελα να σας επισημάνω ένα θέμα το οποίο ανησυχεί πάρα πολύ την Ευρωπαϊκή Δημοκρατία. Το Facebook από την αρχή της εβδομάδας ε, έχει εισαγάγει μια νέα πολιτική διαφήμιση η οποία δυσχεραίνει τη δυνατότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά και των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων να μπορούν να εκπέμπουν διαφημίσεις ε, στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου. Τα τμήματα που αφορούν το Κοινοβούλιο, την Κομισιόν, το Συμβούλιο έχουν στείλει επιστολέ, στον κύριο Νίκ Κλέγκ και διαμαρτύρονται για αυτή τη νέα πρακτική. Μέχρι τώρα όμω το Facebook δεν έχει αντιδράσει. Εγώ πιστεύω ότι είναι παντελώς απαράδεκτο το ότι μία ιδιωτική εταιρεία ε, ξεκινώντα από κάποια γραφεία στι ΗΠΑ να αποφασίζει αυτή η εταιρεία το πώ θα διεξαχθεί η προεκλογική εκστρατεία. Αυτό είναι ίση, είναι απαράδεκτο, το Facebook προσπαθεί να επιβάλλει σε δημοκρατικά εκλεγμένους θεσμούς όπως είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα πολιτικά κόμματα να επιβάλλει πράγματα. Εμείς όμως έχουμε δικαίωμα να ε, κάνουμε προεκλογική εκστρατεία στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αυτό το νέο, τη νέα τους πολιτική δυσχεραίνουν τη δουλειά μας. Καλό λοιπόν τους συναδέλφους να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και προτείνω τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα να συνεργαστούν από κοινού, να στείλουν μια ανοιχτή επιστολή στον κύριο Ζάκαμπακ, να διαμαρτυρηθούν και να ζητήσουν την αμελητή ανάκληση αυτής της πολιτικής. Άλλοι δύο έχουν ζητήσει το λόγο για διαδικαστικό και μετά θα προχωρήσουμε στην ε, διαδικασία στην ψηφορία. Η κυρία Τούνσταν, παρακαλώ, έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, πάρα πολλοί με ρωτάνε γιατί ε, μοίρασα αυτά ε, τα κίτρινα χαρτιά, αύριο θα τα βλέπετε και στους διαδρόμους σας, να τα πήρατε κιόλας. Να ακούσετε το εξής, στις 19 Απριλίου έχουμε την επέτειο ε, της εξέγερσης ε, στη Βαρσοβία του γκέτο. Εμείς στη Βαρσοβία το εορτάζουμε αυτό με αυτά τα κίτρινα μαντήλια. Ε, γι' αυτό λοιπόν ας τα μοιράσουμε την τελευταία ημέρα να είναι ένα σαφές μήνυμα με αυτά τα μαντήλια καρφίτσες ότι εμείς είμαστε εδώ για να μην επιτρέψουμε να επαναληφθεί τέτοιου είδους έγκλημα. Ποτέ πια. Δεν ήταν διαδικαστικό, αλλά τέλος πάντων παρόλα αυτά θεωρώ ότι άξιζε που λάβατε το λόγο. Ε, επόμενος μιλητής για διαδικαστικό και μετά θα προχωρήσουμε ε, στην ψηφοφορία. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Επειδή το θέμα της Ίντερ ε, βγήκε από τη μερίσια διάταξη, για ένα μόνο λεπτό θέλω να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά από 30 χρόνια για τη συνεργασία που είχαμε. Ειδικά όσον αφορά τα εμπορικά θέματα, τα τελευταία χρόνια, τους τελευταίους μήνες ε, πετύχαμε πάρα πολλά. Όταν ξεκίνησα εγώ ήμασταν 12 κράτη, τώρα είμαστε 28. Όταν ξεκίνησα εγώ δεν υπήρχε καν αίθουσα ολομέλειας για μας και τώρα βρισκόμαστε εδώ σε αυτή την αίθουσα. Θα ήθελα να μου επιτρέψετε να ευχαριστώ κυρίως το κρατήδιό μου, την κάτω Σαξονία και τη Γερμανία για το γεγονός ότι ήρθα εγώ εδώ χωρίς να είμαι γεννημένη Γερμανίδα και παρόλα αυτά μου έδωσαν τη δυνατότητα να υπηρετήσω τη Γερμανία για 25 συναπτά έτη. Αυτό είναι γνήσια, αμυγός δημοκρατικό. Αγαπητοί συνάδελφοι, να είμαστε υπερήφανοι για αυτά που μπορέσαμε να επιτύχουμε από κοινού. Ε, σας ευχαριστώ θερμά για όλα και ελπίζω ειλικρινά να υπάρχει και ζωή μετά το Κοινοβούλιο για τους Ευρωβουλευτές. Thank you, let me also... Ευχαριστώ, συνάδελφοι. Και εγώ σας ευχαριστώ και σας εύχομαι ό,τι καλύτερο. Ο κύριος Καθιστάλτο έχει το τελευταίο διαδικαστικό. Μετά θα ψηφίσουμε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ναι, έχω ένα διαδικαστικό για το άρθρο 320, 327. Η ερμηνεία που θα ψηφίσουμε σήμερα είναι πλήρης τροποποίηση του κανονισμού. Πρόκειται για πρόταση που θα εγκριθεί με απλή πλειοψηφία. Αυτό ακριβώς απαιτείται στην ερμηνεία. Είναι η ίδια πρόταση που τροποποιεί τον κανονισμό και που δεν έφτασε σε πλειοψηφία μέχρι τώρα. Το προτινόμενο κείμενο θέτει νέα νομικά ζητήματα που επιδέχονται διαφορετικές ερμηνείες αλλά και διακριτική εκτίμηση Ποιες είναι οι παράμετροι λοιπόν για να καταλήξουμε στον πραγματικό χαρακτήρα που χρειάζεται για να δημιουργείται μια πολιτική ομάδα και τον πολιτικό προσανατολισμό. Ποιο αποφασίζει κατά πόσο τηρούνται οι παράμετροι και τα κριτήρια αυτά, ο πρόεδρο του Κοινοβουλίου μόνο του, με συνένεση στην ε, διάσκεψη των πρόεδρων, με πλειοψηφία, με συνένεση και ποιε είναι οι συνέπειε μια εκτίμηση μη συμμόρφωση. Τέλο, ε, ποια είναι τα μέσα το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς για να αλλάξει μια απόφαση. Υπάρχουνε. Όλα αυτά μένουν ανοιχτά. Στο τέλος της θητείας ξαφνικά βιαζόμαστε και θέλουμε να αλλάξουμε τους κανόνες που διέπουν την ε, δημιουργία πολιτικής ομάδας. Κάτι το οποίο θα αφήσει ανοιχτά πολλά νομικά ζητήματα, αλλά θέτει και σε κίνδυνο τη δημοκρατική λειτουργία του σώματος. Η ψηφοφορία αυτή είναι μια επίθεση στην δημοκρατία και γι' αυτό σας ζητώ μαζί μου να καταψηφίσετε πείτε όχι στην ερμηνεία αυτή και πείτε ναι στη δημοκρατία. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος. Κύριε Καστάλντο, έχουμε ακολουθήσει τους κανόνες της διαδικασίας. Δεν θα αναφερθώ στα σημεία 3 και 4, των 4 με 6. Η συζήτηση έχει γίνει. Δεν θα συζητήσουμε άλλο. Ψηφίζουμε. Πρώτο θέμα στην εμείς διάταξη είναι η ερμηνεία του άρθρου 32, παράγραφος 5, πρώτο εδάφιο, δεύτερη περίπτωση του κανονισμού. Με ονομαστική ψηφοφορία παρακαλώ. Μπορείτε να ψηφίσετε. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τώρα, περνάμε στο επόμενο θέμα. Πρόκειται για την έκθεση Κορό. Πρωτόκολλο στη Συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκή Κοινότητα και του Βασιλείου τη Δανία για τα κριτήρια και μηχανισμού που προσδιορίζουν το κράτο που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτηση ασύλου και σχετικά με το Eurodac. Πάλι με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλο τη ψηφοφορία. Εγκρίθηκε. Επόμενο θέμα. Έκθεση ΝΙΚΑ, θέσπιση του Ορίζον Ευρώπη και τον κανόνων συμμετοχή και διάδοσή του Ψηφίζουμε το σύνολο του κειμένου 203 ε, CP1. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 203 CP2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Άρθρο 3. Παράγραφος 2 σημείο Β. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. Το επόμενο καταπίπτη. Τροπολογία 205 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίφθηκε. Τροπολογία 203 συπ 4 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 207 τώρα διαλατάς ο χειρός υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται 203 CP5 τότε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται το επόμενο καταπίπτει άρθρο 6 208 τροπολογία με ονομαστική ψηφοφορία ψηφίστε παρακαλώ τέλος απορρίφθηκε άρθρο 6 Παράγραφος 7, ονομαστική ψηφοφορία για το 209. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 203 CP6. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Άρθρο 6, παράγραφος 8. Α, όχι, διορθώνει ο πρόεδρος. Συγγνώμη. Θα ψηφίσουμε την τροπολογία 66 CP1. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 203 CP7 D. 66 CP2 D που είναι ίδιες. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 211 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε το 203 CP8 και 71 CP1. Υπέρ παρακαλώ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ετυλογική σκέψη 3, 212 με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος. Απορρίφθηκε. Οπότε ψηφίζουμε την τροπολογία 4 και 203 CP9 υπέρ παρακαλώ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τώρα ψηφίζουμε την πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπής με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος. Εγκρίθηκε. Συγχαρητήρια. Τώρα συνεχίζουμε με την έκθεση του κύριου Έλερ. Πρόγραμμα υλοποίηση του Horizon Ευρώπη. Ονομαστική ψηφοφορία 290. Όχι, με διάταση όρος υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 300, ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος. Απορρίφθηκε. Ψηφίζουμε την πρόταση επιτροπή με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος. Εγκρίθηκε. Περνάμε τώρα στην 309 υπέρ, κατά, ψηφίστε ηλεκτρονικά μάλλον, 301, εγκρίθηκε. Τώρα περνάμε στην έκθεση Ντάντι, εποπτεία της αγοράς και συμμόρφωση των προϊόντων. 214, ονομαστική ψηφοφορία, διορθώνει ο Πρόεδρος. Κύριε Ζόλοβιτ. Κύριε Ζούλο, συγγνώμη, δεν σας δέχετε το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Ζήτησα το λόγο γιατί θέλω να σας πω να ψηφίσετε τις δικές μου τροπολογίες ε, σύμφωνα με το F95 σημείο 3 του κανονισμού η εισαγωγή της υποχρέωσης το να αναφέρεται στην ετικέτα η πρόληψη προϊόντος προστατεύει την υγεία και αποθαρρύνει τον αθέμητο ανταγωνισμό. Είναι αλήθεια ότι η συμφωνία στον τριμερή διόλογο είναι ε, πολύ σημαντική για τη συμμόρφωση του προϊόντος όμως ε, το να το εγκρίνεται αυτό σημαίνει ότι θα ε, καταφερθούμε κατά τις συμφωνίες που έχουμε από το Συμβούλιο. Ε, δεν ε, μπορούμε να έχουμε το Made in. Το Made in είναι προστασία για τους πολίτες, τους εργαζομένους και τις επιχειρήσεις. Πολλές φορές έχει υποστηρίξει το Κοινοβούλιο το Made in και θέλουμε να το κάνει εκ νέου. Ευχαριστούμε. Ο εισηγητής, ο κύριος Δάντη, θέλει το λόγο. Και εσείς ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρέπει να πω ότι εμείς είμαστε κατά του αιτήματος αυτό. Ίσως ο κύριος Τζούλο να μην ήταν παρόν στους τρίμερες διαλόγους και να μην ε, συνειδητοποιεί το πόσο δυσκολευτήκαμε για να πετύχουμε μια τέτοια συμφωνία μετά από τόσα χρόνια που τελικά θα μας επιτρέψει να έχουμε μια αγορά που θα είναι αντικείμενο εποπτείας και όχι μια αγορά όπως σήμερα όπου το 32% των παιχνιδιών δεν, δεν συμμορφώνονται με τους κανόνες και το 40% των ηλεκτρικών ειδών δεν συμμορφούνται με την νομοθεσία. Εμείς εργαστήκαμε σκληρά επί το κειμένου αυτού. Αυτό το κείμενο υπερψηφίστηκε από τον κύριο Τζούλον και από την ομάδα EFTD. Επίσης υπερψηφίστηκε και από την Ιταλική κυβέρνηση στο Συμβούλιο και Αναμένουμε αν ε, τόσο σημαντικό είναι αυτό το θέμα για τον κύριο Τζούλο και το EFTD, ο κανόνας για το Made in ε, μπορεί να το κάνει ακόμη στο κείμενο, στο Συμβούλιο, ζητώντας από τον Υπουργό Ντιμάιο να κάνει αυτά που έπρεπε να γίνουν ε, και αυτά που κάνουμε εμείς στην κυβέρνησή μας. Σας ζητώ λοιπόν να απορρίψετε την πρόταση αυτή. Ευχαριστούμε κύριε Ντάντη. Τώρα ψηφίζουμε την πρόταση του κύριου Ζούλου που είναι να ψηφίσουμε με μονομένα τις τροπολογίες. Δυνατά ισχυρός. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίφθηκε. Οπότε ψηφίζουμε τη 214 με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος. Εγκρίθηκε. Οπότε ολοκλήρωσε την πρώτη ανάγνωσή του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιο. Συγχαρητήρια. Περνάμε στην έκθεση Σαλντεμόζε για την πρόθεση τη δίκαια μεταχείριση και τη διαφάνεια για του επιχειρηματικού χρήστε επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβηση. Ονομαστική ψηφοφορία στην τροπολογία 142. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλο. Εγκρίθηκε. Οπότε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ολοκλήρωσε την πρώτη του ανάγνωση. Συγχαρητήρια. Τώρα περνάμε στην έκθεση Dalton. Καλύτερη επιβολή και εξυγχρονισμό των κανόνων τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την προστασία των καταναλωτών. Ε, παρακαλώ, έχετε το λόγο, κύριε Τονίμεν. Δυστυχώ η οδηγία αυτή δεν λύνει το καυτό ζήτημα της ε, ε, διπλής ποιότητας των ε, προϊόντων. Υπάρχουν ε, διάφορες εξαιρεσει που επιτρέπει να πολλούνται προϊόντα σε ίδια συσκευασία διαφορετικής όμως ποιότητας. Και οι πολίτες έτσι αντιμετωπίζουν η διάκριση σε βάρος τους κάποιοι. Οπότε από 25 χώρες μέλη διάφοροι πολίτες έχουν υπογράψει την τροπολογία η οποία απαγορεύει αυτές τις αθέμητες πρακτικές. Σας ζητώ λοιπόν να υπερψηφίσετε αυτή την ε, τροπολογία. Ευχαριστώ. Υπάρχουν 38 ευρωβουλευτές που ζητούν ε, κάτι τέτοιο. Αυτό το αίτημα. Παρακαλώ. Νομίζω ότι υπάρχουν αρκετοί. Οπότε ψηφίζουμε. Α, και ο κύριος Ντάλτον θέλει το λόγο. Παρακαλώ, για ένα λεπτό. Κύριε Ντάλτον. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κοιτάξτε, Μα πήρε τόσο χρόνο να καταλήξουμε σε συμφωνία. Είναι η τελική συμφωνία στην οποία κατέληξαν όλε οι πολιτικέ ομάδε στον τριμερή διάλογο. Συμφωνήσαμε. Έχουμε νέου κανόνε για αυτήν την διτή ποιότητα. Αντιμετωπίστηκαν όλα τα ζητήματα. Οποιαδήποτε τροπολογία τώρα περάσει θα σκοτώσει το φάκελο ολόκληρο και θα καταστραφεί ένα ολόκληρο κεκτημένο για τους καταναλωτές ε, που μας πήρε τόσο χρόνο να πετύχουμε. Έχουμε μια καλή συμφωνία και θα ήθελα το Κοινοβούλιο να στηρίξει αυτή τη συμφωνία ώστε να γίνει και νομοθεσία όσο γίνεται πιο γρήγορα. Καλώς ψηφίζουμε τότε την πρόταση της κυρίας Τον Σούμεν με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος της ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. Οπότε δεν θα ψηφίσουμε την τροπολογία αυτή, αλλά την 111 με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ για την 111. Τέλος. Εγκρίθηκε. Οπότε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έτσι ολοκλήρωσε την πρώτη του ανάγνωση. Συγχαρητήρια κύριε Ντάλτον και συνεχίζουμε με την έκθεση Αγιούσο διαφάνεια και βιωσιμότητα της αξιολόγησης κινδύνου στην αλυσίδα τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε την τροπολογία 171 με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λοιπόν ολοκλήρωσε την πρώτη ανάγνωση. Συγχαρητήρια στην κυρία Γιούσο. Και τώρα περνάμε στην έκθεση The Grandes Pasquale, συμπληρωματικό πιστοποιητικό προστασίας για τα φάρμακα. Θέλετε το λόγο, παρακαλώ κύριε The Grandes. Δεν επιβεβαίνονται αυτό. Θα προχωρήσουμε λοιπόν στην ψηφοφορία για την προσωρινή συμφωνία, ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται παρακαλώ. Λήξη. Εγκρίνεται. Κύριε Πασκόλτε Γκράντες, θέλετε το λόγο τώρα, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολύ σύντομα. Θέλω να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο για αυτό το αποτέλεσμα. Είμαι σίγουρος ότι θα ωφελήσει την υγεία των Ευρωπαίων πολιτών. Θέλω να ευχαριστήσω τους και συζητητές για την συνεργασία τους και μαζί καταλήξαμε να βρούμε αυτό το συνενετικό αποτέλεσμα. Θέλω να ευχαριστήσω όλο το Κοινοβούλιο γιατί αποχωρώ μετά από 15 χρόνια για την συνεργασία και θέλω να πω σε όλους ε, τους βουλευτές ανεξάρτητα από το σε ποια ομάδα ανήκουν, ήταν τιμή για μένα να είμαι σε αυτό το κοινοβουλίο και να συνεργαστώ μαζί τους. Ε, εγώ ε, ονειρεύτηκα πάντοτε ε, αυτό το είδος στην Ευρώπη και θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες μου όλα αυτά τα χρόνια γιατί πραγματικά με στήριξαν στην εργασία μου. Ευχαριστώ για την πίστη τους, την Άννα, τη Μερσέντες, τη Μακαρένα, την Αλεσάνδρα. Σας ευχαριστώ όλες σας και αντίο. Κύριε Ντεγκράντε Πασκουάλ, και εγώ να σα ευχηθώ κάθε επιτυχία και συγχαρητήρια γιατί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ολοκλήρωσε την πρώτη ανάγνωση για την εκθεσή σα. Τώρα, περνάμε στην έκθεση Σαλίνη, Διαστημικό Πρόγραμμα τη Ένωση και Οργανισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση για το Διαστημικό Πρόγραμμα. Η Επίτροπος θέλει να πάρει το λόγο, παρακαλώ, μέρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ πολύ. Ε, πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό θέμα που καταδεικνύει την πρόθεσή μας να διατηρήσουμε αλλά και να ενισχύσουμε την θέση μας σχετικά με το διάστημα. Ε, πέντε δηλώσεις λοιπόν που αφορούν στην ε, συμμετοχή των κρατών μελών και σε θέματα κυρίως εφαρμοστικών πράξεων, η πρόσβαση στο διάστημα, η σύσταση επιτροπής, η εξέλιξη του Κοπέρνικους. Αυτά τα θέματα, αυτό το κείμενο θα κατατεθεί στις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς προχωράμε λοιπόν στην ψηφοφορία. 2.30 παρακαλώ, υπέρ, κατά. Αποχές, εγκρίνεται. 2.29 με ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη. Απορρίπτεται. Θα περάσουμε τώρα στην ψηφοφορία 228 με ανάταση χειρός, υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Θα ψηφίσουμε τώρα την πρόταση Κομισιόν με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται. Λήξη. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στον κύριο Σελήνη. Περνάμε τώρα στην έκθεση Μλίναρ, πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη για την περίοδο 2021-2027. Η Επίτροπος, παρακαλώ. Παρακαλώ, Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αυτή η ψηφοφορία επιβεβαιώνει τη δεσμεύση να εφαρμόσουμε για πρώτη φορά ε, μια ευρωπαϊκή προσέγγιση για να οικοδομήσουμε ψηφιακέ ικανότητε και οικοδομέ σε στρατηγικού τομεί, όπω παραδείγματο χάρη ε, η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, και η τεχνητή νοημοσύνη και θα υποστηρίξουμε και την ψηφιακή ενιαία αγορά. Η Κομισιόν όμω θέλει να κάνει την εξή δήλωση. Η Κομισιόν δεν μπορεί να συμφωνήσει με τι αλλαγέ ό,τι αφορά ε, τι ε, προσωρινέ μεταφορέ κονδυλίων που δίνονται στα κράτη-μέλη υπό τον ε, κοινό επιμερισμό. Αυτό θέτει προβλήματα συμβατότητα με άλλε νομοθετικέ προτάξει, παραδείγματο χάρη με τον κοινωνισμό περί κοινών διατάξεων. Θέλει να τονίσει η Κομισιόν την ανάγκη να έχουμε μια οριζόντια προσέγγιση στο θέμα αυτό στι διαπραγματεύσει για το επόμενο πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Αυτό τίθεται προ εξέταση από του συνομοθέτε. Σα ευχαριστώ. Θα προχωρήσουμε στην ψηφοφορία με ανάταση χειρό. 206 τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές. Αγκρίνεται και θα ψηφίσουμε την πρόταση της Κομισιόν με ονομαστική ψηφοφορία. άρχιτη ψηφοφορία. Λήξη. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια, κυρία Μλίναρ. Προχωράμε στην έκθεση γκίγκολτ Πρόγραμμα φισκάλης για τη συνεργασία στον τομέα της φορολογίας. Ψηφίζουμε την τροπολογία 4 το κείμενο στο σύνολό του, έτσι όπως έχει υποβληθεί από την Επιτροπή. Με ένα θεσχυρός, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και θα ψηφίσουμε την πρώτη της Κομισιόν με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Να περάσουμε τώρα στην έκθεση Herbrandi, πρόγραμμα για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα, live. Και η Επίτροπος Πιερκόφσκα θέλει πάλι το λόγο. Παρακαλώ, ευχαριστώ πολύ. Αυτή η νομοθετική πρόταση είναι πολύ επίκαιρη. Έρχεται σε μια στιγμή Οπότε οι Ευρωπαίοι πολίτε και ιδίω οι νέοι διαμαρτύρονται, βγαίνουν στου δρόμου και ζητούν να κάνουμε περισσότερα για το κλίμα και για το περιβάλλον. Είναι ένα παρακαλώ μήνυμα για να ε, συμφωνήσουν τα θεσμικά όργανα. Τρει δηλώσει θέλουν να κάνει η Κομισιόν. Λοιπόν, την Κομισιόν που οι συνομοθέτε αποφάσισαν να διατηρήσουν το λογότυπο του LIFE, γιατί αυτό δεν σέβεται την οριζόντια προσέγγιση, να μην έχουμε συγκεκριμένα λογότυπα για τα προγράμματα. Με τον πολιτικό προπολογισμό δεύτερον, η Κομισιόν θεωρεί ότι υπάρχει έλλειψη αιτιολόγηση για την διαδικασία εξέταση ε, για τη ρήτρα τη μη γνωμοδότηση. Τρίτον, η Κομισιόν επιβεβαιώνει ότι η ανοιχτή διάρκεια του προγράμματο είναι υπό την επιφύλαξη στο προνόμιο τη Κομισιόν να παρουσιάσει ένα πρόγραμμα που το live για το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό ε, πλαίσιο. Όλα αυτά είναι προς εξέταση από τους συνομοθέτες. Ε, λοιπόν, Περνάμε στην τροπολογία 105 CP1 με ένα τεσχυρό υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 108 με ονομαστική ψηφοφορία άρχεται. Λήξη. Απορρίπτεται. Θα περάσουμε λοιπόν στην τροπολογία 41 με ένα τασιχυρός υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 109 με ένα τασιχυρός υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Δηλαδή θα περάσουμε στην τροπολογία 42 με ένα τασιχυρός υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 110 με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται. Λήξη. Απορρίπτεται. Τροπολογία 111 με ονομαστική. Άρχεται. Λήξη. Απορρίπτεται. Τροπολογία 112 με ανάταση χειρός υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 105 συμπι 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 113 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 51CP υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 105CP5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 106 τροπολογία με ονομαστική ψηφορία άρχεται. Λήξη. Απορρίπτεται. 107 με ονομαστική άρχεται. Λήξη. Απορρίπτεται. Επομένω, περνάμε στην πρόταση Κομισιόν στο σημερινό τη με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται ψηφοφορία. Λήξη. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στον κύριο Χερμπράντι. Επόμενο. Έκθεση Βιέντεν Χόλτσερ και Χαουτάλα, πρόγραμμα δικαιοσύνη. Τροπολογία 78 CP1 με ανάταση χειρό. υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 78 CP2 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 78 CP3 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 78 CP4 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 78 CP5 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 78 CP6 σε δύο μέρη, με ένα τασιχυρό. Για το πρώτο τμήμα, υπέρ, κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα την πρόταση τη Κομισιόν με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται. Λήξη. Εγκρίνεται. Συνάδελφοι, από την τελευταία έκθεση, τελευταία φορά πρόεδρε από τι ψηφορίε, ε, θα ήθελα λοιπόν εκφράσω την εκτιμησή μου για τα τελευταία δύο χρόνια για τη συνεργασία μας και θα ήθελα να ευχηθώ κάθε επιτυχία σε όσους συμμετέχουν στις εκλογές και στους υπόλοιπους που δεν συμμετέχουν κάθε επιτυχία για τα υπόλοιπα. Ευχαριστώ συνάδελφοι. Για σας ε, είναι το χειροκρότημα. Περνάμε τώρα στην έκθεση της κυρίας Βαλέρο, πρόγραμμα δικαιώματα και αξίες, τροπολογία 116 με ονομαστική. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη. Απορρίπτεται το κείμενο στο σύνολό του. 115 τροπολογία υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τώρα ψηφίζουμε την πρόταση της Κομισιόν με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται. Λήξη. Εγκρίνεται. Τώρα, έχουμε μια σειρά διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπιών. Έχουμε ένα σημείο για το θέμα αυτό οι κοινοβουλευτικέ αντιπροσωπείε, αντιπροσωπείε στι Βρυκτέ Κοινοβουλευτικέ Επιτροπέ, αντιπροσωπείε στι Επιτροπέ Κοινοβουλευτική Συνεργασία και στι Πολυμερεί Κοινοβουλευτικέ Συνελεύσει. Έχουμε πρόταση για απόφαση από τη διάσκεψη των Προέδρων και το αρχικό κείμενο. Μανάτα χειρό, υπέ. Απλώ να πω για την παράγραφο 1, σημείο Β, γραμμή 5, το αρχικό κείμενο. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Έτσι λοιπόν έρχεται η ψηφοφορία για τον έλεγχο, λήξη. Εγκρίνεται. Έτσι λοιπόν τώρα θα ψηφίσουμε την πρόταση για απόφαση υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Σας ευχαριστώ συνάδελφοι και σε λίγο θα περάσουμε στις επεξηγήσεις ψήφου. Όσοι δεν συμμετέχετε λοιπόν, παρακαλώ να αποχωρήσετε ησύχως. Συνάδελφοι, για άλλη μια φορά σας παρακαλώ να αποχωρήσετε ησύχως για να προχωρήσουμε στις αιτιολογήσεις ψήφου και να δείξουμε ε, σεβασμό σε όσους θα συμμετάσχουν στη διαδικασία αυτή. Θα ξεκινήσουμε σε λιγότερο από ένα λεπτό. Λοιπόν, για άλλη μια φορά ευχαριστούμε όλους όσοι φεύγουν και βγαίνουν από την αίθουσα. Ε, προχωράμε στις αιτιολογήσεις ψήφου. Πρώτη έκθεση της ε, κυρίας Ντανίκα σχετικά με το πρόγραμμα Ορίζων, καθορισμός ε, κανόνων συμμετοχής. Πρώτος που έχει δει στο λόγο είναι η κυρία Μάιερ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Μάιερ. Μισό λεπτό για άλλη μια φορά σας παρακαλώ να βγείτε από την αίθουσα για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στις αιτιολογήσεις ψήφου. Κυρία Μάγια, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η ε, αφέμαξη, η διαρροή εγκεφάλων, το brain drain, ε, αυτό είναι εκτεταμένο με βάση το Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ και στην περίπτωση αυτή η χρηματοδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι καθοριστική σημασία για να διευκολύνει την διεθνή συνεργασία. Το πρόγραμμα Horizon 2020 σημαίνει ότι οι επιστήμονες ε, είναι πολύ σημαντικές ε, μπαταρίες θα λέγαμε γιατί μπορούν να εξερευνήσουν θέματα τεχνολογίας. Σήμερα λοιπόν συζητήσαμε για το διάδοχο πρόγραμμα από το 21 στο 27. Θεωρώ ότι όλα αυτά βέβαια είναι αρκετά μακριά για τη Βρετανική κυβέρνηση που μοιάζει να λειτουργεί μόνο από ώρα σε ώρα αλλά στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να παραμείνουμε μέσα στο πρόγραμμα αυτό. Η δική μας η φήμη είναι ότι επιδιώκουμε τη ρηξικέλευτη έρευνα, αλλά ξέρουμε ότι η φήμη πάρα πολύ εύκολα ή το καλό όνομα πολύ δύσκολα αποκτάται και πολύ εύκολα χάνεται. Ο κύριος Πάλμερ, ε, η χρηματοδότηση του προγράμματος Ορίζων είναι πολύ δύσκολη στη δική μου την περιοχή. Έχουμε κονδύλια που περικόπτονται για την έρευνα. Περίπου 7 εκατομμύρια όμως έχουν δοθεί για να στηριχθούν επιχειρήσεις. Αυτή η χρηματοδότηση ε, σε όλα αυτά τα χρόνια και για πάρα πολλές γενιές ε, δεν είναι σωστή. Έχουμε όμως άλλα κοινωνικά κοινωνικά προγράμματα τα οποία θα έπρεπε να στηριχθούν. Η Βρετανική κυβέρνηση πρέπει λοιπόν να αντικαταστήσει την πολιτική οτιδήποτε λιγότερο δεν είναι αποδεκτό. Εάν υπάρχουν αυτά τα χρήματα για το Brexit και αν υπάρχουν και τα χρήματα για να αντικατασταθούν τα ευρωπαϊκά προγράμματα με τη λύρα, οτιδήποτε λιγότερο είναι απαράδεκτο. Εμείς ε, όλες οι περιοχές ε, της δικής μου της περιφέρειας θα πρέπει να την χάνουν τις δίκες μεταχείρισης και ακριβώς αυτό ζητάμε. Ο κύριος Ντέβα, για ένα λεπτό. Το Horizon 2020 είναι ένα από τα προγράμματα τα πιο πετυχημένα όλα αυτά τα χρόνια. Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι η έρευνα πρέπει να βρίσκεται στην καρδιά και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του κόσμου γιατί παράγει πρωτότυπη έρευνα. Θέλω ιδιαίτερα να ευχαριστήσω τη Σούσαν Κέρκ, Μπεν Άλμερ, Αντριάλεν, Ντάνιελ Χάμελτον, Ίγκριτ Γκρότολ, Λιγκάι, Λεβερ Κάβιαρ, Άλμπον Αντώνιον, Κέβιν Ρόμπινσον και Ντάνιελ Χόλουερτ. Διότι όλοι έχουν κάνει τη διαφορά στο έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στη συνεργασία τους μαζί μου. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Ντέβα. Επόμενος ο κύριος Σένφελτ. Ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Πρόεδρε, το πρόγραμμα Ορίζον Ευρώπη και μόνο από το όνομά του είναι καταπληκτικό. Είναι πολύ καλό το όνομα αυτό γιατί ακριβώ δείχνει ποιοι είναι οι στόχοι μα. Δηλαδή θέλουμε μια σύγχρονη Ευρώπη, μια ανταγωνιστική Ευρώπη στι παγκόσμιε αγορέ και θέλουμε μια Ευρώπη που να βασίζεται στην καινοτομία. Και ακριβώ γι' αυτό το πρόγραμμα, κατά τη γνώμη μου, αξίζει την πλήρη υποστήριξή μα. Και εδώ δεν πρόκειται μόνο για στήριξη των 84 εκατομμυρίων που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλουμε 120. Θέλω εδώ να αναφερθώ σε κάποιο ωφέλη του προγράμματος, που είναι και πολλά. Πρώτα απ' όλα, εδώ υπογραμμίζουμε την σημασία που έχουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις με 70% στις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δεύτερον, οι διαφορές ε, που υπάρχουν πρέπει να καλυφθούν. Είναι αλήθεια ότι στην Ευρώπη υπάρχουν χώρες που διαθέτουν τεράστια κονδύλια για την έρευνα και άλλες όχι. Ευχαριστούμε πολύ που μου δίνετε το λόγο, λέει ο κύριος Αχραντήλ. Πραγματικά είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένο που η τελευταία φορά που παίρνω το λόγο εδώ, ε, στο σώμα, ε, με κάνουν να είμαι θετικός. Άλλες προηγούμενες φορές ήμουν επικριτικός, επέκρινα διάφορες νομοθετικές πράξεις που υιοθετούσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όμως γι' αυτό το πρόγραμμα, το Horizon, είναι ακριβώ πρόγραμμα σαν αυτά τα οποία πρέπει πάντα να στηρίζουμε υπέρ της έρευνας, της καινοτομίας, της επιστήμης. Οπότε είμαι ιδιαίτερα ευτυχής, συμφωνώ με το πρόγραμμα αυτό και ελπίζω να έχουμε μια φιλόδοξη συμφωνία και φιλόδοξη χρηματοδότηση. Επιτρέψτε μου επίσης να πω ότι μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ελπίζω να ενταχθεί στο πρόγραμμα αυτό το Ηνωμένο Βασίλειο παρόλα αυτά, γιατί είναι ένα στενό εταίρο μα στην επιστήμη και την έρευνα. Ο κύριο Ποσπισίλ, παρακαλώ, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ με ικανοποίηση υποστήριξα αυτή τη συμφωνία, γιατί κάθε ευρώ που επενδύουμε στην έρευνα είναι ένα ευρώ που περνάτε καλά. Χαίρομαι λοιπόν που έχουμε μια προσωρινή συμφωνία και χαίρομαι που βλέπω ότι τα ποσά που θα επενδυθούν έχουν αυξηθεί. Επίσης, με χαρά σημειώνω ότι η ροή χρημάτων είναι μεγαλύτερη και θα υπάρξουν λοιπόν περισσότερες επενδύσεις ε, για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, για τις τεχνολογίες της υγείας και σε άλλους πολύ σημαντικούς κλάδους. Αν η Ευρώπη θέλει να ε, συναγωνιστεί με τους άλλους εταίρους παγκοσμίω, ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε αυτή το πολύ σημαντική ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Ο κ. Καπούτο, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Στον νέο κανονισμό Horizon Ευρώπη έχουμε το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Έρευνας που είναι το πιο φιλόδοξο. Είναι σημαντικό μήνυμα το να δίνουμε το 35% της χρηματοδότησης ε, στις τεχνολογίες που σέβονται το κλίμα. 35 δισεκατομμύρια ευρώ στα 120 για την ε, περίοδο 2021-2027. Επίσης, έχουμε ε, ξεκάθαρους στόχους όπως η μείωση των εκπομπών του άνθρακα στις πόλεις και θα επικεντρωθεί το πρόγραμμα στους στόχους θεμάτες. Επίσης, έχουμε την νέα αναφορά ε, προκειμένου από το εργαστήριο να έχουμε στην αγορά τεχνολογίες υψηλής δυναμικής και να βοηθήσουμε τις ε, καινοτόμες επιχειρήσεις να αναπτύξουν τις δέστος. Το μόνο αρνητικό είναι ότι δεν έχουν αποκλειστεί από τη χρηματοδότηση τα ορυκτά καύσιμα και ε, πιθανότατα όμως θα ήταν κάτι που θα έπρεπε να κάνουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, κύριος Κώστα για ένα λεπτό. Συγγνώμη και πάλι. Φυσικά σας γνωρίζω πολύ καλά, αλλά διάβαζα την, τον κατάλογο. Κυρία Κώστα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλή αυτή η είδηση. Ε, έστω και μια μερική συμφωνία για το πρόγραμμα Horizon 2020 ε, με όλα αυτά τα δισεκατομμύρια που θα δώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ελπίζω βέβαια να γίνει σεβαστή η συμφωνία γιατί βασίζεται στην ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χαίρομαι πάρα πολύ για δύο κυρίως θέματα. Μπορέσαμε δηλαδή να πετύχουμε να ενταχθεί ε, το θέμα το κοινωνικό σε όλο το θέμα που αφορά την βιομηχανική πολιτική. Θα ήταν περίεργο αυτό να μην υπάρχει από κοινού με την επιστημονική έρευνα και σε διάφορα θέματα. Το δεύτερο που πετύχαμε, και αυτό είναι ένα σημαντικό δικό μας επίτευγμα, το να υπάρχει ένα κλάστερ θεματικό που θα έχει τον τίτλο ε, «Πολιτισμό σε 2,5 δισεκατομμύρια θα είναι επιδότηση για την έρευνα και 300 εκατομμύρια για το νέο Cloud Cultural Heritage». Το το οποίο αντιμετωπίζει την ε, πρόκληση στο, στην ε, κληρονομιά μας, στην πολιτιστική κληρονομιά μας. Όλα αυτά ενισχύουν τις ευρωπαϊκές προσπάθειες. Χάναν, για ένα λεπτό. Ε, κύριε Πρόεδρε, πότε θα επικρατήσει αυτή η άποψη ότι η πολιτική και τα στελέχη ε, είναι καλύτερο να, ε, και πιο κατάλληλοι να αποφασίζουν για το πού θα διοχετεύονται τα χρήματα για την έρευνα. Εγώ προηγούμενα, πριν γίνω πολιτικό, ήμουν δημοσιογράφο και πραγματικά πρέπει να σα πω ότι κανένα από όσα επιδοτήθηκαν δεν απέδωσε. Οι μεγάλε τομέ, αυτά που άλλαξαν την ζωή των ανθρώπων στην Αμερική και αλλού, Κανένα από αυτά δεν χρηματοδοτήθηκε από κυβέρνηση. Ε, όπως και αυτοί που επέφεραν την βιομηχανική επανάσταση. Είμαστε εδώ λοιπόν σε δύσκολη θέση, ζητάμε αυτούς που θα είναι οι αποδέκτες. Ε, βεβαίως ε, είναι μια πολύ καλή ιδέα, αλλά νομίζω ότι όταν είναι περιορισμένος ο προπολογισμό, αυτή είναι και η βέλτιστη δυνατή λύση. Βεβαίως και εγώ θέλω να δαπανάμε χρήματα για την παιδεία, αλλά όταν ακούω κάποιους που προτείνουν ότι το μέγεθος μετράται με το, η επιτυχία με συγχωρείτε με το μέγεθος του προπολογισμού, δεν είμαι σίγουρος ε, κατά πόσον ε, τα καταφέραμε καλά. Ε, τώρα, το επόμενο πρόγραμμα του κυρίου Κρίστιαν Έλε, ο κύριος Χάναν και πάλι για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αυτή είναι η τελευταία μου ομιλία στην Ολομέλεια και θα ήθελα να δράξω την ευκαιρία να ευχαριστώ εσάς, το ε, προσωπικό, τους ε, διερμηνείς, τους συνεργάτες και θέλω να σας πω, ε, στενοχωριέμαι πάρα πολύ που δύο χρόνια μετά τις εκλογές όπου το 85% των πολιτικών επέστρεψαν, τώρα βρισκόμαστε σε ε, άλλη μια περίπτωση που θα έχουμε εκλογές. Περνάμε τώρα στις επεξηγήσεις ψήφου για την έκθεση του κυρίου Νίκολα Ντάντη εποπτεία τη αγοράς και συμμόρφωση των προϊόντων. Μία μιλήτρια, η κυρία Μίτση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. για τους καταναλωτές. Όταν αγοράζουν καινούργια προϊόντα, καλλιντικά για παράδειγμα, ε, πρέπει να ξέρουν ότι αγοράζουν ασφαλή προϊόντα. Δεν συμβαίνει όμως αυτό πάντα, γιατί πολλές φορές προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά είναι επικίνδυνα. Τα μόνα προϊόντα που πρέπει να βρίσκονται στην αγορά πρέπει να είναι τα ασφαλή προϊόντα. Γι' αυτό λοιπόν και χρειαζόμαστε κανόνες, έλεγχο, συμμόρφωση. και για τους παραγωγούς, αυτοί οι οποίοι συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές, να ξέρουμε ποιοι είναι. Χρειάζεται ευρωπαϊκή νομοθεσία που να προστατεύει τους καταναλωτές όταν αγοράζουν προϊόντα που μπορεί να είναι επικίνδυνοι. Σήμερα υπερψήφισα την ε, νομοθεσία αυτή γιατί βελτιώνει ακριβώς την ασφάλεια των προϊόντων για τους καταναλωτές έτσι ώστε να υπάρχει περισσότερη δικαιοσύνη στην αγορά μας. Οι κανόνες αυτές θα προστατεύουν ακόμα περισσότερο την υγεία των καταναλωτών. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Έκθεση Ντάλτον ε, τώρα όσον αφορά την καλύτερη επιβολή και εξυγχρονισμό των κανόνων για την προστασία των καταναλωτών. Παρακαλώ. Ο κύριος Πάλμερ, ευχαριστώ. Είναι άδικο όταν δεν μπορεί να αγοράσει κανείς κάτι το οποίο πραγματικά να αξίζει τα χρήματα. Όμως γίνονται τις τιμές. Γι' αυτό και χρειάζεται έλεγχος στις χώρες μέλη και χαίρομαι για όσου έχουν κάνει εκστρατεία στο Ηνωμένο Βασίλειο, για παράδειγμα. Χρειάζεται και συντονισμένη αντίδραση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα με ε, μέτρα τα οποία να ελέγχουν την κατάσταση σε διάφορες αλυσίδες όπως είναι το Google. Υπάρχουν ε, διάφορα αποτελέσματα τα οποία εμφανίζονται στο Google όταν κανείς ψάξει και αμέσως θα βρει τα ίδια. Ζητάω λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να το αντιμετωπίσει αυτό και τα κονδύλια τα οποία κυκλοφορούν στην Ευρώπη να δίνονται και να κατανέμονται πιο δίκαια. Ευχαριστούμε ο κύριος Πόσπισιλ. Ευχαριστώ. Αφού δίστασα για καιρό υποστήριξα τελικά την πρόταση αυτή, η οποία δεν είναι τέλεια σε ό,τι αφορά την καταπολεμήση της δυτής ποιότητας στα τρόφιμα. Μία ε, τροπολογία που δεν πέρασε καταπολεμούσε την ε, δυτή ποιότητα. Δυστυχώς δεν πέρασε η τροπολογία αυτή και λυπάμαι. Έτσι λοιπόν, ο συμβασμός στον οποίο καταλήξαμε είναι ένα μισό βήμα εμείς ως Τσεχική Δημοκρατία και άλλα κρατεμέλη έχουμε προϊόντα της ίδιας ποιότητας και με την ίδια ονομασία. Βέβαια δεν αρκεί η συμβαστική πρόταση και ελπίζω ότι στο μέλλον το νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Κομισιόν θα αντιμετωπίσει το θέμα αυτό και αν πράγματι δούμε ότι δεν αρκεί ο συμβιβασμός, τότε στο μέλλον θα υιοθετήσουμε κάτι παραπάνω. Η επόμενη έκθεση είναι μια έκθεση της κυρίας Αγιούσο, διαφάνεια και βεσιμότητα της αξιολόγησης κινδύνου στην αλυσίδα τροφίμων στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρακαλώ, Σοσνιέρς, για ένα λεπτό. Οι πιστοποίησεις ε, των ε, προϊόντων ουσιαστικά προέρχονται όταν έχουμε την έγκριση από τους αρμόδιους φορείς. όμως ε, κανένας ποτέ δεν ε, έχει πει ότι μπορούμε να δράσουμε κατά μιας απόφασης ενός τέτοιου οργανισμού. Δεν έχει νόημα λοιπόν. Και υπάρχουν ε, κάποιοι άνθρωποι που κάνουν έρευνα για το τι μπορούμε ή δεν μπορούμε να τρώμε. Αυτή η οδηγία επίσης είναι πάρα πολύ γενικόλογη και εδώ απλώς βλέπουμε ότι όλα θα έπρεπε να γίνουν εγκαίρως. Όμως δεν μεταφράζεται σε συγκεκριμένα μέτρα και γι' αυτό καταψήφισα την έκθεση αυτή. Τελευταία έκθεση για την οποία έχουμε επεξήγηση ψήφου είναι η έκθεση του κυρίου Γκράντας Πασκάλ για τα πιστοποιητικά σχετικά με τα ιατρικά προϊόντα. Η κυρία Φαρία για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ε, πρόεδρε, σήμερα το 60% των φαρμάκων είναι γενώσιμα που παράγονται από ευρωπαϊκές εταιρείες και φαίνεται ότι αυτή η αγορά ε, φέρνει περισσότερες ευκαιρίες και εξοικονομήσεις για το σύστημα υγείας. Εγώ υπερψήφισα την έκθεση αυτή γιατί πιστεύω ότι αυτή η εξαίρεση ε, θα είναι θεμελιώδες έτσι ώστε ε, να έχουμε ποιοτικά γενώσιμα για τους Ευρωπαίους πολίτες και θα αυξήσουμε την προσφορά στην Ευρώπη προκειμένου να έχουμε ασφάλεια εφοδιασμού στην αγορά και να μειώσουμε και τις ελλείψεις. Επίσης, θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε τα τρίτα κράτη, να εξάγουμε σε τρίτα κράτη προϊόντα που θα έχουν παραχθεί ε, με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες. Το CCP είναι μία επέκταση ε, στο δίπλωμα ευαισθητεχνίας και πρέπει να πούμε ότι κανένα κεκτημένο δικαίωμα δεν θα ζημιωθεί με αυτό τον κανονισμό θα πρέπει να διατηρηθεί η Ενωμένη Ευρωπαϊκή Ένωση σε έναν κόσμο συνεχούς ανταγωνισμού και θα πρέπει να προωθήσουμε αυτή την ευρωπαϊκή βιομηχανία που προωθεί την ευρωπαϊκή οικονομία. Κύριο Καπούτο, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο νέο κανονισμό, όσον αφορά το συμπληρωματικό πιστοποιητικό προστασία για τα φάρμακα που μόλι εγκρίναμε θα δώσει τη δυνατότητα στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων να διευρύνει τι αρμοδιότητε του και κατά αυτόν τον τρόπο θα δημιουργηθούν νέε θέσει εργασία. Αυτή τη στιγμή θα έχουμε μια πολιτική πολύ πιο βιώσιμη. Ας μην ξεχνάμε ότι οι φαρμακοβιομηχανίε αντιμετωπίζουν πολύ έντονο ανταγωνισμό εξαιτία των εταιριών των επιχειρήσεων από τι τρίτε χώρε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να υπάρχουν πολύ δεσμευτικοί κανόνε όσον αφορά τη διάθεση φαρμάκων στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή τη στιγμή θα καταφέρουμε να προωθήσουμε γενώσιμα φάρμακα τα οποία θα φέρουν αυτό το σπληρωματικό πιστοποιητικό προστασίας και θα μπορούμε κατά αυτόν τον τρόπο να εξάγουμε με ασφάλεια τα φάρμακα αυτά και στην αγορά εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πέρα από όλα αυτά τα ωφέλη θεωρώ ότι όλος ο κλάδος της φαρακομαβιομηχανία θα μπορούσε να υποφεληθεί. Ας μην ξεχνάμε ότι πολύ συχνά ξεχνάμε στον τομέα αυτό τους πολλού διαφορετικού κανόνες που υπάρχουν για την προστασία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνία. Σας ευχαριστούμε κύριε Καπούτο. Συνεχίζεται η συνεδρίασή μας στις 3 το μεσημέρι.